Αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι 9 και 10. Θα ξεκινήσουμε την κοινή αυτή ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή ΔΕΒΕ και Επιτροπή ΙΝΤΕ για την ε, για το νέο κανονισμό σε σχέση με την υλοτόμηση και τους δασικούς πόρους. και τον ε, ε Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΔΕΒΕ, τον κύριο Ερίχε Γκρέο Γκρέο-Σάλλον. Καλημέρα σε όλους σας. Επιτέλους έχουμε μια μέρα με ήλιο στις Βρυξέλλες. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι πιο πολύ Ιταλική και Ισπανική μέρα και όχι Βελική μέρα. Είναι προφανώς θυσία να είμαστε σε 9 το πρωί εδώ, αλλά αξίζει τον κόπο αυτή η θυσία. Το κάνουμε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όχι μόνο το περιβάλλον, <clears throat> αλλά και τα στοιχεία αυτά του περιβάλλοντος που διατηρούν μια μορφή ζωής πολλών ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εργάζονται για την προστασία των ε, δασών και τη χρήση των πόρων που έρχονται από τα δάση. Ζητά συγγνώμη η πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης, η Βίντα Μακάβελ, ως Βρετανή καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μας. Επίσης, με την ευκαιρία <clears throat> θέλω να πω και εγώ ορισμένα λόγια για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Παρά του το γεγονός ότι εδώ και πολύ καιρό έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, ιδίω μέσω του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των νόμων, την διακυβέρνηση και τα θέματα του Διεθνούς Εμπορίου Δασικών Πόρων στα αγγλικά, το ακρόνιμο είναι FLECT. Τώρα, αν το προφέρω καλά, βέβαια, και επίσης. Οι συμφωνίες αυτές καλύπτουν τα θέματα εμπορίου ξύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ισχύουν από το 2013. Όλες αυτές οι διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις έχουν επιτρέψει με κάποιο τρόπο να μειωθεί η παράνομη υλοτόμηση και το παράνομο εμπόριο ξύλου, αλλά δεν έχουν εμποδίσει αυτή η παράνομη υλοτόμηση να συνεχιστεί σε ορισμένες χρονικές στιγμές και αυτό εξαρτάται φυσικά από την χρονική συγκύρια και σε ορισμένε περιπτώσει αυξάνεται η παράνομη υλοτόμηση. Όπω καταλαβαίνετε, αυτή δεν είναι μόνο μια πρακτική που βλάπτει το περιβάλλον, αλλά αλλάζει και τις συνθήκες διαβίωσης των πληθυσμών που ζουν σε δασικές εκτάσεις. Η Επιτροπή Ανάπτυξης λοιπόν έχει αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στις συμφωνίες <clears throat> σύνδεσης σε εθελοντικό επίπεδο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιων χωρών που παράγουν ε, ξυλία στην Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική με θετικά κίνητρα αφενός αλλά συγχρόνως προσπαθώντας και να βοηθήσουν τον αγώνα κατά της διαφθοράς, την ε, αποδυνάμωση του κράτους δικαίου Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μερικές, σε μερικές περιπτώσεις κράτη που έχουν αστοχήσει και επομένως δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την παράνομη υλοτόμηση. Οι συμφωνίες λοιπόν που έχουν επιτευχθεί έχουν δώσει μια θετική όθηση σε μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει μέσα στις χώρες αυτές. Αλλά η εφαρμογή αυτών των συμφωνιών ή δεν έχει επιτευχθεί ακόμα ή έχει τελματωθεί σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό για πολλούς ε, λόγους, πάνω απ' όλα, επειδή δεν υπάρχει απαραίτητη πολιτική πίεση, αλλά συγχρόνως και επειδή υπάρχει και κενό διακυβέρνηση σε πολλές από αυτές τις χώρες και έλλειψη ικανότητα για να μπορέσουν να ε, χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν οι αρρωγές που δίδονται σε χρηματικό επίπεδο. Υπάρχουν και ορισμένε χώρες και ιδίως η Ινδονησία που έχουν προχωρήσει πολύ στον έλεγχο της παράνομης υλοτόμησης. Το Ελεκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσφατα δημοσίευσε μια έκθεση όπου αναφέρει και ορισμένα κενά στην εφαρμογή αυτών των συμφωνιών που οδηγούν και σε χορήγηση βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ελεκτικό Συνέδριο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει και ένα σχέδιο εργασίας πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες αυτές με σαφέστερους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και ένας ειδικό προϋπολογισμός για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Εμείς από την Επιτροπή Ανάπτυξης πιστεύουμε ότι πράγματι θα πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση προσθέτων πόρων, θα πρέπει να ελέγξουμε με ένα πιο συνεπή και συνεχή τρόπο την χρήση αυτών των πόρων και την ε, επιζήτηση των στόχων που θέλουμε να έχουμε. Πιστεύω ότι και η σημερινή συνεδρίαση που περιλαμβάνει τρεις επιτροπές, Ιντα, Τέβε και Χένβι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να πούμε ιδέες για το πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υποδεικνύει και επίσης και πώς θα αξιολογήσουμε το σχέδιο δράσης FLEGT και πώς θα προχωρήσουμε και σε μεταρρύθμιση της ε, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοτομία είναι ένα στοιχείο που έχει πολλές πτυχές, έχει να κάνει και με τη σταθερότητα σε πολιτικό επίπεδο πολλών από τις εμπλεκόμενες χώρες, έχει να κάνει μια άλλη πτυχή με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά σε τελική ανάλυση η πιο σημαντική πτυχή είναι αυτή που έχει να κάνει με το να διατηρηθεί ο χώρος στον οποίο ζουν και εργάζονται όλοι αυτοί οι οποίοι εξαρτώνται από τα δάση και την υλοτομία. Ευχαριστώ και θα δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Ίντα για να έχουμε και την άποψη της τρίτης επιτροπής που εμπλέκεται σε αυτή τη συνέντευξη. <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόφανως η στρατηγική του να υπάρχει εμπόριο το οποίο βασίζεται στην ε, παραγωγή προσθέμενης αξίας είναι πολύ σημαντικό και στο θέμα της ξυλίας και το θέμα της ε, βιώσιμης δασοκομείας και γι' αυτό είμαστε πάντα πρότιμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να βελτιώσουμε την κατάσταση που παρουσίασε ο Ενρίκε. 12 χρόνια μετά τη διατύπωση του σχεδίου FLECT δεν υπάρχει ακόμα σύστημα αδειοδότησης και ελπίζω ότι τώρα θα ξεκινήσουμε με την ιδιοδότηση αυτή για την ε, Ινδονησία, να εφαρμοστεί το σχέδιο αδειοδότησης στην Ινδονησία. Και θα είναι ίσως το πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να δούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο στους δύο τομείς που συνδέονται με την ε, δασοκομεία. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε <clears throat> ότι υπάρχουν οι απαραίτητε συνθήκε για να διατηρηθεί η ποιότητα του περιβάλλοντο και τη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Χθε συζητήσαμε για τα θέματα των ορεικτών που προέρχονται από ζώνες εμπόλεμες. Είναι η ίδια λοιπόν ακριβώ προβληματική. Θα πρέπει να δούμε όλη την αλυσίδα προσθέμενη αξία για τα προϊόντα αυτά αυτή πρέπει να είναι η πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για όλα αυτά τα νομοθετήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ξεκινούμε με τις παρουσιάσεις. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λορέντσο από την DG DevCo. Ευχαριστώ πολύ. Εάν θέλετε μπορούμε να αρχίσουμε την παρουσίαση με τις διαφάνειες. On the screen? It's not on the screen. Okay, good morning. Um Καλημέρα σας, λέει η κυρία από την Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτή η κοινή συνεδρίαση είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, ούτως ώστε να τα πούμε, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις για το σχέδιο δράσης, να δούμε τώρα αυτές τις διαφάνειες προεισαγωγικά, ούτως ώστε να φρεσκάρουμε την μνήμη μας για το περί τίνος πρόκειται κατόπιν της ε, αξιολόγησης. Όπως όλοι γνωρίζετε, το σχέδιο δράσης FLEGT ξεκίνησε το 2003 για να καταπολεμήσουμε την παράνομη υλοτόμηση και το σχετιζόμενο εμπόριο. Ήταν διεφέκτο τότε για την ε, Διεύθυνση ε, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Είναι κοινή προσπάθεια και βέβαια και και τα κράτη-μέλη και συνεργαζόμενες χώρες. Εδώ πέρα είναι διπλός ο στόχος. Πρώτα-πρώτα ε, είναι εμπορική συμφωνία, ε, αλλά υπάρχει και η πτυχή διακυβέρνηση. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν ε, διάφορες δυσκολίες ακριβώς λόγω του διτού διπλού στόχου. Δηλαδή με λίγα λόγια πρόκειται για ένα περίπλοκο εργαλείο και όχι κάτι το παραδοσιακό ως πρόγραμμα. Είναι ένα πακέτο πολιτικής και ρυθμιστικών μέτρων. Ε, υπάρχουν 7 άξονες που καλύπτει αυτό το σχέδιο δράσης ή πρόγραμμα δράσης ε, διακυβέρνηση όσον αφορά τη συμμετοχή του δυτικού τομέα, την χρηματοδότηση, τις επενδύσεις και καλύπτεται και η κοινωτική νομοθεσία. τα βασικά στοιχεία αλλά και επιτεύγματα αυτού του προγράμματος. Αναφέρεται στην αρχή ακριβώς ότι έχουμε αυτό το VPA, δηλαδή αυτού του είδους την εκούσια συμφωνία συνεργασίας του 2005 και έτσι δόθηκε εντολή διαπραγματευτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε αυτή η συμφωνία συνεργασίας είναι το επίκεντρο αυτού του προγράμματος δράσης, ούτως ώστε να ρυθμιστεί το θέμα της εξαγωγής και υπάρχουν κάποια πιστοποιημένα προϊόντα υλοτομίας, επίσης παρέχεται άδεια πρόσβαση στην αγορά και με αυτές τις συμφωνίες επίσης θα έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση αυτές τις χώρες, θα έχουμε καλύτερη υποχρεωσή λογοδοσίας, διαφάνεια, εμπλοκή όλων των ε, ενδιαφερομένων. Τώρα, άλλος άξονας αυτού του προγράμματος είναι συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Δεν θα πει και ο συναδελφός από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Τώρα, η αξιολόγηση του προγράμματος. Ήρθε η ώρα της μετά από 11 χρόνια κατά τα οποία τρέχει το πρόγραμμα. Αυτό ήταν επιταγή του νόμου, αλλά θεωρήσαμε ότι με δεδομένες τις αλλαγές της συγκυρίας είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν. Αξιολογούμε πάνω στις επιδόσεις του προγράμματος και τους 7 άξονες του προγράμματος και είναι αναπόσπαστα συσχετιζόμενο με τους ελέγχους του ελεγκτικού συνεδρίου υπάρχει συντονισμός με τη διαδικασία αξιολόγησης του κανονισμού για την υλοτομία. Πρόσφατα προέγυψαν αυτά. Ακόμα βρίσκεται να εξελίξη αυτή η διαδικασία που θα καταλήξει σε κάποια έκθεση. Ε, έκθεση του Μαΐου τέλος πάντων σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά και η αξιολόγηση έχει ως μειονέκτημα το ότι έχει κάποια όρια όσον αφορά τα δεδομένα. Τα δεδομένα για την εμπορία αλλά και τα επιτεύγματα σε επίπεδο διακυβέρνησης. Τώρα, μεθοδολογία και επιτέμοντας τα άλλα μέτωπα, καλύτερη νομοθεσία. Έχουμε τη Διευθύνουσα Επιτροπή, τα κρατημέλη. Τώρα, πριν το τα υπέρ και τα κατά, σε σχέση με την αξιολόγηση, πρέπει να πούμε ότι ήταν δύσκολη αυτή η διαδικασία, γιατί το πρώτο που μπορεί να πει κανείς για το FLEGT είναι αυτό που αναφέρθηκε πριν αρχίσει η παρουσίαση, δηλαδή η αδειοδότηση. Και θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι το FLEGT είναι ιδιαζόντως περίπλοκο. Άρα με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε το εξής. Αυτές οι εγκρίσεις, οι άδειε ε, ήταν το πιο απλό στοιχείο, αλλά εκεί δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Εδώ δεν μπορούμε ότι είναι επίτευγμα. Τα ελληθή επιτεύγματα όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση για την δασοπονία είναι κάτι το οποίο δεν έχει μετρηθεί. Επομένως έχουμε αυτά τα επιτεύγματα, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι απτά τα αποτελέσματα. Να δούμε τώρα. Ποια είναι τα θετικά του Φλέγκτ. Πρόκειται για κάτι καινοτόμο. Είναι επίσης ε, κάτι πάρα πολύ επίκαιρο, κάτι το οποίο υποστηρίζει ο ιδιωτικός τομέας ε, κοινωνικών πολιτών, όλοι οι εμπλεκόμενοι οι οποίοι σχετίστηκαν με αυτή τη διαδρομή και Υπάρχει καλή σχέση κόστους ε, αποτελέσματος. Και πρόκειται για κάτι το οποίο έδωσε τη προστιθεμένη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν μόχλευση στην αγορά, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής. Και έτσι επιφέραμε μεταβολές στην διακυβέρνηση. Οπότε υπήρξε ωφέλεια κατόπιν συντονισμού των κρατών μελών. Τώρα σε επίπεδο επιτυχιών του ΦΛΕΚΤ έχουμε 15 χώρες, 6 συμφωνίες συνεργασίας που είναι στη φάση της ε, υλοποίησης και άλλες 9 ε, που τώρα είναι στη δικασία διαπραγμάτευσης και ελπίζουμε ότι το FLEGT θα επιδράσει και στα όσα γίνονται στην Ινδονησία. μεγάλη μας επιτυχία αυτή όσον αφορά ε, ε, τα προϊόντα υλοτομίας τα οποία έχουν τύχη αδειοδότησης και θα εξαχθούν κατά τα τέλη του ενεστώτος έτους. Τώρα θα σας πει κι άλλα η συνάδελφος αλλά η επιτυχία συνεχίστηκε και όσον αφορά την πολιτική για τους κρατικούς διαγωνισμούς. Σαφώς και αυτό είχε επίδραση στην αγορά. Και παγκοσμίω πολλοί μας μιμήθηκαν. Χώρες που καταναλώνουν τέτοια προϊόντα όπως η Αυστραλία και η Ιαπωνία τέτοιες χώρες άρχισαν να θεσπίζουν μέτρα κατά της παρανομισύλλοτομίας, άρχισε ο διμερής διάλογος και ε, με την μεγαλύτερη αγορά που είναι η Κίνα. Οπότε θα έχουμε η ανάπτυξη τέτοιων πολιτικών για τις ε, προμήθειες και αυτά φυσικά και θα επηρεάσουν την ε, αγορά στις περισσότερες χώρες. Τώρα, τα μειονεκτήματα του Φλέκτ, όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση. Αναφέρθηκε προηγουμένως το ότι δεν είναι τόσο στεγανός ο προγραμματισμός σε επίπεδο επιτροπής και κρατών μελών. αυτές οι συμφωνίες συνεργασίας είναι περίπλοκες, ε, χαρακτηρίζονται από ένταση αξιοποίησης των πόρων και το θέμα είναι ότι όσον αφορά τη διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη η επιρροή των νομοθετημάτων που θεσπίζονται. Οπότε ε, πρέπει να υπάρξει περισσότερη προσοχή όσον αφορά την χρηματοδότηση και τις επενδύσεις που δεν έχουν φτάσει σε επίπεδο που ήταν επιθυμητό. Οπότε βλέπουμε βέβαια ότι και τελευταία δεκαετία άλλαξε πάρα πολύ η συγκυρία και το περιβάλλον και ε, τώρα για την καταστροφή των δασών έχει αλλάξει η κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τις μεταβολές στην παγκόσμια αγορά. Συστάσεις τώρα. Η εταιρεία συμβούλων που έκανε την αξιολόγηση ε, μιλά για το ότι θα πρέπει ψυχογραφική βάση και θεματική βάση να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και άρα να υπάρχει ad σχεδιασμός των ε, μέτρων και δράσεων να αντιμετωπίσουν την ερήμωση για το των δασών, κάτι το οποίο βέβαια είναι γενικότερο θέμα. Και θα πρέπει να δούμε τι πολιτικές θα διαμορφωθούν. Και επίσης να συνδυαστούν αυτά με πρωτοβουλίες για να υπάρχει συμπληρωματικότητα. Το έγγραφο εργασία από την υπηρεσία δεν έχει ακόμη προκύψει. Ε, τέλη Ιουνίου θα το έχουμε. Αυτό το έγγραφο ε, κυρίως ασχολείται με την αξιολόγηση και όχι με το μέλλον. Γίνεται εκεί κάποια συνοπτική παρουσίαση. Δεν χαράζει καινούργιες πολιτικές. Είπαμε πρώτα να υπάρξει στην υπηρεσία προβληματισμός και κατόπιν να προγραμματίσουμε. Μας είπαμε ότι το FLEGT ε, αποδίδει καλή σχέση κόστους αποτελέσματος, είναι δόκιμο για την επίτευξη του σκοπού που θέλουμε και επομένως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, τα προβλήματα της αναποτελεσματικότητας τα προβλήματα στον κακό ή μέτριο ε, συντονισμό. Τώρα, τον Ιούνιο είπαμε ότι πρόκειται να εγκριθεί αυτό το έγγραφο εργασίας της υπηρεσίας και είπαμε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή που έρχεται επί Ολλανδικής Προεδρίας. συντονισμο ε, τωρα τον ιουνιο ειπαμε οτι προκειται να εγκριθει αυτο το εγγραφο εργασιας της υπηρεσιας και ειπαμε οτι θα ολοκληρωθει αυτη η διαδρομη που ερχεται επι προεδριας ειχαμε και τα, το, το, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, οπότε επί τη βάση της αξιολόγησης θα γίνει μια ευρύτερη αξιολόγηση ούτω ώστε να μπορούμε να δούμε τι επιλογές υπάρχουν και να αντιμετωπίσουμε την καταστροφή και περίμεση των δασών. Thank you very much. And now... ευχαριστούμε και τώρα μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Άντλη από τη ΓΑΜΑ Περιβάλλον ο οποίος θα μας δώσει μια διαφορετική οπτική γωνία για το σχέδιο δράση Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας, αξιότιμοι προβλευτές και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και εμένα τη δυνατότητα να κάνω αυτή την παρουσίαση. Σε σχέση με την παρουσίαση της συναδέλφου από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΤΕΦΚΟ, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι ε, δεν ε, χρειάζεται νομίζω να σας πείσουμε για το πόσο πολύπλοκο είναι αυτός ο κλάδος ε, και πόσο τεράστια είναι η μετάβαση που προσπαθούμε να επιφέρουμε σε πολλές από τις χώρες με τις οποίες ε, συνεργαζόμαστε έχουμε πει ότι είναι πολύπλοκη πολιτική κατάσταση. Μιλήσαμε για την ε, Ινδονησία, ένα ομοσπονδιακό κράτος με πολύ διαφορετικές απόψεις ανάλογα με την περιοχή της χώρας. Το να τα φέρεις κοντά όλα αυτά είναι δύσκολο. Σίγουρα σημειώνουμε πρόοδο στην Ινδονησία τώρα, αλλά αντιμετωπίσαμε δυσκολίες. Αν σας τα έλεγα αυτά πριν από έξι μήνες, θα σας έλεγα ότι όλα είναι μετέωρα, γιατί τελευταία στιγμή ο Υπουργός Εμπορίου εισήγαγε για, τις, ε, για την επιπλοπία μια τεράστια παρέκκληση. Και πριν από δέκα μέρες εγκρίναμε την κατεξοδότηση πράξη για να εγκρίνουμε τις άδειες στην Ινδονησία σε σχέση με τη διαδικασία μη ένσταση, Δηλαδή ελπίζουμε δεν θα υπάρξει ένσταση. Και αν γίνει έτσι θα τεθεί σε ισχύ στα μέσα Αυγούστου. Οπότε και η τρίμηνη διαδικασία με τα κράτη-μέλη θα ξεκινήσει για τη δημιουργία των απαιτούμενων διοικητικών δομών και αν όλα πάνε καλά πριν τα τέλη του έτους θα έχουμε ε, το πρώτο φορτίο ε, ξυλό από την Τονισία στην Ευρώπη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και από πλευράς φλέκτα τα ωφέλη ε, που θα αποκομίσει και η ίδια η Ινδονησία μετά τη σκληρή δουλειά που έκανε με αυτό το σύστημα θα τους δώσει πλέον εκτήματα. Και άλλες χώρες που το σκέφτονται και διερωτώνται κατά πόσο να ακολουθήσουν την πορεία αυτή ή όχι θα δουν αυτά τα ωφέλη και ελπίζουμε το Ινδονησιακό σύστημα να είναι ένας καταλήτης για να έχουμε περαιτέρω πρόοδο και στο μέλλον. Τώρα έρχομαι στον κανονισμό για το ξύλο, για τα προϊόντα υλοτομίας. και θα ήθελα να κάνω λόγο για τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις του κανονισμού. Το δεύτερο είναι η αξιολόγηση και το τρίτο είναι η υλοποίηση, η εφαρμογή. Τι κάνει αυτός ο κανονισμός λοιπόν για τα προεντελειοτομίες. Απαιτεί ε, την δέωση επιμέλεια από τους διαφόρους φορείς. Θα πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουν ότι το ξύλο ή τα προεντελειοτομίες που αγοράζουν ε, και διαθέτουν στο εμπόριο στα κράτη-μέλη της Ένωσης προέρχεται από νόμιμες πηγές. Είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε κινδύνους, risk-based, δεν υπάρχει έλεγχο στην είσοδο των χωρών. Υπάρχει υποχρέωση του φορέα, και αυτή την υποχρέωση πρέπει να την ελέγχουν τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια απαγόρευση, δηλαδή δεν μπορεί να διατεθεί ε, στο επόριο παράνομο ξύλο και ο κανονισμός έχει κυρώσεις. Οι αρμόδιοι φορείς ε, ελέγχουν την ε, εφαρμογή και αν ανακαλύψουν ότι δεν έχει εφαρμοστεί αυτή η υποχρέωση, επιβάλλουν κυρώσεις. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει απόδειξη ιχνηλασιμότητας Είδαμε και από την εξελόγηση ότι υπήρξαν καθυστερήσεις. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ε, μια διαφορετική διοικητική ε, διαδικασία και δομή και μέθοδο εργασίας που σημαίνει ότι θα πρέπει να ορίσουν οι ειδικοί αρχή σε κάθε χώρα, θα πρέπει να θεσπίσουν αυτές τις ποινές, τα πρόστιμα. Απαιτεί επίσης ε, τη δημιουργία ενός συστήματος για τον έλεγχο των φορών, όχι 100% έλεγχο, αλλά όπως είπαμε βάσει της προσέγγισης αυτής, risk-based. Και όπως είπα, δεν ελέγχονται ε, στην είσοδο, ε, άρα δεν έχουμε ένα τελωνιακό ε, ούτως σύστημα. Και ο ρόλος ε, των κρατών είναι να ελέγχουν όλα αυτά και εμεί θα ελέγχουμε αν εφαρμόζουν σωστά τα σχετικά τα κράτη-μέλη. Τώρα έρχομαι στην αξιολόγηση. Βασιστήκαμε σε εκθέσεις από τα κράτη-μέλη, στο input από τις δημόσιες διαβουλεύσεις που είχαμε και είχαμε επίσης και άμεσες επαφές με πολλούς ε, διαφορομένους φορείς και έτσι καταλήξαμε στην αναφορά που σας παρουσιάσαμε πρόσφατα. Στην αναφορά μας αυτή λέμε ότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως ο κανονισμός έχει τις δυνατότητες να επηρεάσει τα μάλα καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας. Ε, βέβαια, οι πολλοί ενδιαφέρομενοι φορείς ε, αναγνωρίζουν το αληθές αυτή της δήλωση και οι διεθνείς προσπάθειες είναι σημαντικές. Αναγνωρίζεται αυτό. Αναγνωρίζουμε όμως επίσης ότι απαιτούνται από τα κράτη-μέλη και από τον ιδιωτικό τομέα περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή και επίτευξη των στόχων του κανονισμού. Με βάση τα στοιχεία λοιπόν αποδεικνύονται σε πολλά κράτη-μέλη αρμόδιες αρχές. Δεν διέθεταν επαρκείς πόρους για την επιβόλη της νομοθεσίας. Γνωρίζουμε τώρα ότι στα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, γίνονται έλεγχοι στις δημόσιες δαπάνες και από τη στιγμή που βρισκόμαστε στη φάση του ρονταρίσματος τώρα, είναι δύσκολο να τηρηθούν οι νέες υποχρεώσεις ε, για να δοθούν περισσότεροι πόροι εκεί που χρειάζονται ίσως αλλού να δοθούν. Αλλά βλέπουμε σταδιακά να υπάρχει πρόοδος και σε αυτό το τομέα. Οι ευρωπαϊκοί φορείς πλέον λαμβάνουν το μήνυμα ότι πρέπει να πάρουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την νομιμότητα των προμηθειών τους. Βέβαια, η έκθεση δείχνει, όπως είπα, ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες από τους αρμόδιους φορείς και τις αρχές για να υπάρχει πλήρης εφαρμογή του κανονισμού. Ρόλος της Κομισιόν είναι να προωθήσει τη συνεργασία και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν επικοινωνίε εκστρατείε για να αυξήσουμε την αισθητοποίηση ε, στην κοινή γνώμη και στους φορείς και ένα από τα θετικά αποτελέσματα. Είδαμε ότι τον κανονισμό τώρα τον εξετάζουν και άλλοι ε, σε άλλα κράτη, παραδείγματος χάρη Αυστραλία. Βλέπουμε θεσπίζει παρόμοια νομοθεσία. Μελετά το θέμα η Ελβετία. Κάποιες αναδυόμενες οικονομίες επίσης αρχίζουν να το εξετάζουν αυτό το θέμα και στην Ιαπωνία που, συνεδρίασε, ε, που συνεδρίασαν Υπουργοί Περιβάλλοντος ε, του G7 ο Βέλε ζήτησε να το δουν και άλλες χώρες και ενδεχομένω να θεσπίσουν αντίστοιχα μέτρα. Όπως είπαμε, ελπίζουμε ότι ο κανονισμός αυτός θα δώσει κίνητρα σε χώρες με τις αθελούς αυτές τις συμφωνίες VPA να προχωρήσουν ε, σε ένα σύστημα αντίστοιχο με αυτό της συντονισίας που αν εφαρμοστεί η εισαγωγή από την Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζουν τον κανονισμό για τις άδειε και τα λοιπά. Θα πληρούνται όλες οι απαιτήσει για την νομιμότητα του ξύλου. Ωστόσο, προέκυψε ένα ζήτημα στο πλαίσιο της αναθεώρησης, το εξής. Στον κανονισμό για την ε, υλοτομία έχουμε επαρκές πεδίο προϊόντων εύρος επαρκές υπάρχουν κάποιες ασυνέπειες, αυτό διαπιστώθηκε, πίνακες παραδείγματο χάρη. Μάλλον ε, τα τραπέζια, αλλά όχι καρέκλες. Περιλαμβάνω, τα τραπέζια, όχι καρέκλες. Άρα ε, πρέπει να το δούμε. Μήπως πρέπει να επεκταθεί το πεδίο. Τα τελευταία δύο χρόνια και συνεχίζουμε και τώρα έχουμε μια ε, συνεργασία με τα κράτη-μέλη, έχουμε την Επιτροπή ΦΛΕ και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, για να έχουμε ανταλλαγή εμπειριών και να μάθουμε ένα από τον άλλον, ώστε να έχουμε ε, κατευθυντήριε γραμμέ, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κτλ. Και αν θέλετε, αυτή είναι η ήπια πλευρά ε, της προσέγγιση μα Υπάρχει και μια πιο αυστηρή, που είναι η επιβολή η εφαρμογή της νομοθεσίας. Στρέφουμε το 2014. Τότε τι γινόταν είχαμε 18 κράτη-μέλη ακόμη που δεν είχαν σε επαρκή πρόοδο σε τέφα συμμόρφωση. Τον Ιούνιο πέρυσι, τέσσερα μόνο ήταν τα κράτη-μέλη που δεν είχαν ακόμη συστήσει τους ε, απαιτούμενους φορείς, ε, τις ε, απαιτούμενες αρχές και συνεχίζουμε το διάλογο μας με αυτές τις χώρες. Το έχουμε χαλαρώσει λίγο το θέμα βέβαια ε, και εάν ε, τα κράτη-μέλη δεν προχωρήσουν, αυτά τα τέσσερα, θα ξεκινήσουμε και διαδικασίες επί παραβάση. Βέβαια, οι υποσχέσεις που λαμβάνουν, όπως από την Ισπανία, εκεί λήφθη μια απόφαση να μην υπάρχει μόνο μία αρμόδια αρχή, αλλά σε κάθε περιφέρεια να υπάρχει μία αρχή. Αυτό μας δυσκολεύει λίγο τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων αναγνωρίζονται οι ευθύνε που υπάρχουν, ε, ξέρουμε ποιο είναι και το σύστημα διακυβέρνηση στην Ισπανία και περιμένουμε και τα ονόματα ε, των ε, αρχών ανάλογα με την αυτόνομη περιφέρεια μέχρι το τέλος του μήνα. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι, δεχόμαστε ότι απομένουν να γίνουν ακόμη πολλά. Έχουμε την ήπια προσέγγιση που την κάνουμε λίγο τώρα πιο αυστηρή και αυτό δίδει καρπούς και ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μεγαλύτερη πρόοδο. Εγώ, παραδείγματο χάρη, θεωρώ πολύ θετικό το ότι σε κάποια κράτη-μέλη που υπάρχουν καλά συστήματα ελέγχων, ένας από τους δείκτες, μπορεί να είναι αρνητικός δείκτης, είναι ο αριθμός ε, δικαστικών υποθέσεων. Και βλέπουμε να γίνονται δίκες και να επιβάλλονται πρόστιμα. Στον ετήσιο διάλογο με την Κίνα, οι συνάδελφοί μας έδωσαν το μήνυμα στους Κινέζους. Τους είπαμε ορίστε έτσι έχουν τα πράγματα και σημειώστε το πρέπει να δίνετε καλέ πληροφορίε στου οικονομικού σα εταίρου από την Ένωση. Αλλιώ μπορεί να επηρεαστούν οι εμπορικέ σα σχέσει με την Ένωση. Προχωρούν λοιπόν τα πράγματα. Φυσικά και δεν θα πω ότι είναι τέλειο το σύστημα. Πολλά απομένουν να γίνουν. Υπάρχει όμω η δέσμευση. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σα ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο, για τι εξηγήσει που δώσατε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα. Ο κύριο Ζαντό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είχα την ευκαιρία να είμαι εισηγητή στο παρελθόν στην Επιτροπή Ίντα για ορισμένε από τι εθελοντικέ συμφωνίε στα πλαίσια του ΦΛΕΚΤ. Κάναμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό σε μεγάλο βάθο. Νομίζω το 2014, στο τέλος τη της θητεία συγκεκριμένα, συζητήσαμε για την κατεξουσιοδότηση πράξη που αφορούσε την Ινδονησία. Είναι σημαντική αυτή η συζήτηση με κάποιες εντάσεις, γιατί εδώ και κάποια χρόνια όλες οι αξιολογήσεις δείχνανε ότι ένα μεγάλο μέρος των ε, δασικών προϊόντων από την Ινδονησία ε, υλοτομούντο με παράνομο τρόπο. Και δεν υπήρξαν δεν υπήρχαν κατάλληλε δομέ ελέγχου. Βέβαια, έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια η κυβέρνηση της Ινδονησίας ώστε να βελτιώσει την φήμη τη κάτι το οποίο ήταν προφανές ότι έπρεπε να γίνει, αλλά επίση έκανε και μια μεγάλη προσπάθεια εξυγίανση του δασικού τομέα. Αυτό μας παραπέμπει σε όλη τη σημασία και τη φιλοσοφία του ΦΛΕΚΤ. Εμεί ω πράσινοι έχουμε υποστηρίξει αυτό το μηχανισμό από την αρχή, γιατί αποτελεί ένα εργαλείο για να γίνει πιο θεμητό το εμπόριο, πιο δίκαιο το εμπόριο στα προϊόντα αυτά. όπως ελέγχθηκε από την Κομισιόν, είναι το ΦΛΕΚ και ένα εργαλείο για την προστασία των δασικών πόρων, ακόμα και αν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της αποψήλωσης αφορά την μετατροπή των δασών σε αγροτικές γέες. Αλλά είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο δημοκρατικοποίησης της κοινωνίας στα μέρη όπου ε, λειτουργεί το ΦΛΕΚΤ. Δημοκρατία δεν σημαίνει μονάχα βέβαια τις εκλογές και το κράτος δικαίου, αλλά η δημοκρατία <clears throat> αποτελεί και την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, ιδίως των εμπλεκομένων από την κοινωνία των πολιτών, σε όλες τις ε, αλυσίδες παραγωγής, ε, όταν πρόκειται για εξόριξη ή εκμετάλλευση φυσικών πόρων, όπου πολλές φορές σοβή η διαφθορά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το φλέγ και στις περισσότερες χώρες όπου υπάρχουν αυτές οι εθελοντικές εταιρικέ συμφωνίες οι ΜΚΟ πολλές φορές έχουν δείξει την ικανοποίησή τους για αυτή τη διαδικασία. Τώρα βέβαια βλέπουμε ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. το Φλεκτ υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια αλλά δεν υπάρχει ακόμα διοδότηση Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους. Ότι αυτή, αυτός ο μηχανισμός δεν έχει οδηγήσει σε ένα μηχανισμό αντιοδότησης που θα έδινε νόημα σε, όλη αυτή την, σε όλο αυτό το εγχείρημα. Επομένως υπάρχει πίεση να υπάρξουν αποτελέσματα, αλλά εκεί εμφυλοχωρεί ο κίνδυνος του να έχουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν <clears throat> αποτελέσματα βεβαιασμένης εξέτασης. Αν οι πρώτες άδειε δείξουν ότι δεν έχουν απόλυτη σαφήνεια σε ό,τι αφορά την <clears throat> νομιμότητα των προϊόντων ξυλίας που θα έρθουν στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα τεθεί αναφιβόλο όλο το σύστημα. Η ομάδα μου προφανώς υποστηρίζει την πρόοδο που έχει γίνει στην Ινδονησία για τα θέματα αυτά Συγχρόνως όμως πρέπει να είμαστε συλλογικά πάρα πολύ επάγρυπνοι και προσεκτικοί τα πρώτα αυτά προϊόντα που θα έρθουν με αδειοδότηση να μην συνδέονται με υποψίες παράνομης ε, υλοτόμησης, διαφθοράς, μη ανεξαρτησίας των αρμοδίων φορέων, έλλειψη ε, διαφάνειας. Ξέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της ξυλίας παντού και ιδιαίτερα στην Ινδονησία και επομένως εν κατακλείδη είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε αυτή την εταιρική σχέση μεταξύ όλων των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εμπλέκονται αλλά και με την Κομισιόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί <clears throat> ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι πρώτες άδειες που θα εκδοθούν να είναι άψογου χαρακτήρα και θα έχουν υποδειγματικό χαρακτήρα για τις άλλες χώρες και όχι να είναι ένα αντιπαράδειγμα το οποίο θα οδηγήσει σε τελμάτωση της δυναμικής. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπίλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εμείς ε, χαιρετίζουμε ιδιαίτερα αυτήν την ε, απόφαση της Κομισιόν να υπάρξει τροποποίηση στην ε, ρύθμιση για την υλοτομία. Εμείς έχουμε μία ιστορικά πολύμορφη διαχείριση για τους δασικούς πόρους στα κράτη-μέλη μας και φυσικά δεν υπάρχει πάντα συγκρισιμότητα μεταξύ των συστημάτων αυτών. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ταχύτητα η εφαρμογή αυτών των κανόνων. Κατά την άποψή μας θα ήταν ίσως <clears throat> πρόωρο να ζητάμε μια ομοιόμορφη ε, εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Και μέσα στα κράτη-μέλη έχουμε ακόμα την ανάγκη να συνεχίσουμε τις ε, διαδικασίες διαβούλευσης και πληροφόρησης των εμπλεκομένων στην αγορά και φυσικά να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία ώστε να μην υπάρξει μεγαλύτερο γραφειοκρατικό άχθος. Βλέποντας και το, το παράτημα, Πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για το περιεχόμενό του, αλλά νομίζω ότι αν κάνουμε και μία ιδιαίτερη αντιμετώπιση για τις περιοχές αυτές από τις οποίες ε, εισάγονται δασικά προϊόντα, μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την ισότητα ανταγωνισμού και την αηφορία της ευρωπαϊκής υλοτομίας. Ξέρουμε ότι και μέσα στην Ευρώπη χρησιμοποιούμε μόνο 65% των βασικών μας πόρων Επομένω, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πόρο, ένα πολύ σημαντικό πόρο, τον οποίο δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και να εξετάσουμε αν κάποια προϊόντα όπως είναι ο φελός, που είναι κυρίως εισαγόμενο προϊόν, να μπορέσουμε να τον <clears throat> αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο σε εσωτερικό επίπεδο στην Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να μειώσουμε την παράνομη υλοτόμηση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Ο κύριος Χιέλμαρ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολλές φορές είναι σαν τα χρυσόψαρα σε ό,τι αφορά τον οριζόντα μνήμης τους γιατί εργαζόμαστε για πάρα πολλά πράγματα, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε τα προηγούμενα. Εγώ υπήρξα εισηγητής για τον κανονισμό της ε, υλοτόμησης. Αυτό ήταν πριν από κάποια χρόνια. Ε, συγγνώμη, συγχωρήστε με αν δεν έχω στο μυαλό μου όλες τις λεπτομέρειες. Είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ καλό να ξέρουμε ότι υπάρχει τώρα μια συνολική άποψη της εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα και να συνδέσω αυτό το ερώτημα με το συγκεκριμένο, το ευρύτερο θέμα. Το ερώτημα μου το εξή. Ξέρουμε ότι ο κανονισμό για την υλοτόμηση περιλαμβάνει κάποιε κυρώσει. Αυτό ήταν αντικείμενο μεγάλων συζητήσεων όταν γινόταν διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν όμω κάποιε κυρώσει που προβλέπονται από αυτόν τον κανονισμό. Θα ήθελα να ξέρω. Υπήρξε ποτέ κάποιο πέναλτι που να εφαρμοστεί Υπήρξε κάποτε κάποια εταιρεία ή κάποιο άτομο που θεωρήθηκε ότι παραβιάζει αυτόν τον κανονισμό και επομένως επισύρει κάποιες κυρώσεις για αυτόν τον λόγο. Αν η απάντηση είναι όχι, υπάρχουν δύο τρόποι να το δούμε. Θα πούνε κάποιοι συνάδελφοι, μα αυτό δεν είναι καλή εφαρμογή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα για να εφαρμόζεται καλύτερα ο κανονισμός. Μπορεί να υπάρχει και μια άλλη πτυχή που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη προτού Ε, καταλήξουμε σε μια ευρύτερη αντιμετώπιση. Ίσως μπορεί να υπάρχει ενώπιό μας μια πραγματική πρόκληση για να φτάσουμε στο ύψος <clears throat> αυτού του κανονισμού. Και συγγνώμη αν ξεχνά μερικά πράγματα, θα πρέπει να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα δασικά αυτά είδη, <clears throat> η χώρα προέλευσης, όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο. Αυτό καλύπτει πολλά πράγματα, όπως παραγωγής χάρη την ε, χαρτοβιομηχανία. Αν έχετε ένα, ένα εργοστάσιο παραγωγής χαρτομάζας στη Φιλανδία, που πολλές φορές έχει και ξυλία και από την Φιλανδία και από τη Ρωσία που εισάγεται, πώς θα μπορείς κανείς να ξεχωρίσει τις διάφορες πηγές, πώς μπορεί να ξέρει ότι η παραγωγή αυτή γίνεται με το ένα ή το άλλο είδος ε, ε Για να μπορεί κανείς να πει ακριβώς από ποιο δέντρο προέρχεται, η ξυλία αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Είπανε πολλοί οι οποίοι είπαν ότι θα μπορέσει θα μεγάλες εταιρείε να το λύσουν. Η ΑΚΕΑ στη Σουηδία είπε ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και ίσως είναι η πιο κατάλληλη εταιρεία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, αλλά είναι δυνατόν για τις μικρότερες εταιρείες να πούν ότι αυτό το ε, κομμάτι δέντρου ή αυτό το ροκανίδι προέρχεται από το τάδε δασικό είδος και την τάδε χώρα. Έχουμε την ανάγκη φυσικά να διευρύνουμε την εμβέλεια αυτού του νομοθετήματος, γιατί έχουμε νέα προϊόντα, όπως είναι τα πλαστικά που έρχονται από την, από την κυταρίνη των ε, δασικών προϊόντων. Συγχρόνως όμως <clears throat> υπάρχει ένα πρόβλημα να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τα προϊόντα αυτά. Υπάρχει στα σουηδικά αυτό που λέμε γκρουτ, που είναι τα υπολείμματα που μένουν όταν ε, πράγματι έχουμε υλοτομήσει κάποιο δέντρο. Έχει μια μεγάλη αξία αυτό το υπόλοιμα αλλά αν είναι τόσο μεγάλη γραφειοκρατία για να μπορέσει κανείς να εξασφαλίσει ότι αυτό το τελευταίο μέρος του κορμού με τις ρίζες που έχει μείνει θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνουμε αυτά τα νέα προϊόντα, τα οποία πολλές φορές θα είναι πιο πολύπλοκα και θα βασίζονται σε πολλαπλές πηγές. Θα ήθελα να ξέρω την άποψη της Κομισιόν. Θα μπορούσε το πρόβλημα της ε, εφαρμογής αντικείμενο, είναι αποτέλεσμα της τεράστιας πολυπλοκότητας και της δυσκολίας να εφαρμοστούν όλα αυτά και δεν είναι μόνο θέμα θέληση και πόρων. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε διάφορε πρωτοβουλίε που έχουν να κάνουν με την διαφάνεια και την υποχρέωση λογοδοσία για αυτό το τομέα και για όλε τι ανανεώσιμε ε, πηγέ ενέργεια και ενεργειακού πόρου όπως το ETI και άλλες. Οπότε αυτό που πρέπει να γίνει είναι κάτι να κάνουμε όσον αφορά τους ανανεώσιμους ε, πόρους και να εξασφαλίσουμε επίσης βιώσιμη και διάφανη διαχείριση. Ακριβώς και αυτό θα γίνεται και τώρα όσον αφορά τον ε, κανονισμό για την υλοτόμηση και την πρωτοβουλία του το πρόγραμμα τέλος πάντων. Άρα να θεσπιστεί κάτι πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό επί τη βάση των όσων έχουμε πετύχει με τη Συμφωνία Συνεργασίας και το ΦΛΕΚΤ και τον κανονισμό. Θεωρώ ότι τώρα τα καλά, θα υπάρξει ένα πρόγραμμα δράσης για την απερίμωση και υποψήλωση των δασών, οπότε κάτι μπορούμε να πετύχουμε, ούτω ώστε να πάμε στην επόμενη φάση. Έχω όμως δύο-τρεις ερωτησούλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ασχοληθεί περισσότερο για να άρει κάποια προβλήματα ασυνέπειες που υπάρχουν και έτσι να είμαστε πιο συνεπείς στην πολιτική μας για να πετύχουμε τους στόχους μας σχετικούς με το θεματολόγιο 2030. Αλλά βέβαια και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δει όλα αυτά τα θέματα ευρύτερα. Δεύτερη ερώτηση. Ακούσαμε σε σχέση με την αξιολόγηση του κανονισμού ότι μπορεί να υπάρξει διεύρυνση της βεντάλιας των σχετικών προϊόντων. Η μετατροπή των δασών, λέγεται, είναι κίνητρο για παράνομη υλοτομία που οδηγεί στην απερίμωση από ψήλους των δασών. Άρα τι θα γίνει, θα υπάρξει διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή τη ύλη που καλύπτει ο οργανισμό. Τέλο πάντων, είπαμε επίση, σαν τρίτη ερώτηση, ότι στο ΦΛΕΚ δεν μετέχει αρκετά ο ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει μήπω περίπτωση να έχουμε κάποια εργαλεία, κάποια μέσα, ούτω ώστε να έχουμε κάποιο είδου μηχανισμού ε, προαιρετική, υποχρεωτική ρύθμιση, ούτω ώστε να υπάρξει συνεργασία και ταυτόχρονα υποχρέωση ε, λογοδοσίας για την, το τι γίνονται τα προϊόντα από την υλοτομία μέχρι τον καταναλωτή και επίσης να δούμε τι θα γίνει με τον κανονισμό με, για τα ορυκτά και δεν είναι εδώ μόνο το θέμα της σύγκρουσης των νομοθετημάτων αλλά είναι και το κατά πόσο είναι βιώσιμη ε, η αυτή αλυσίδα προϊόντων που προέρχονται από τα δάση. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν τώρα έχει αρχίσει να χαράσει ένα καινούργιο πρόγραμμα δράσης για την ε, αποψήλωση των δασών. Αυτό πώς θα γίνει, θα γίνει με τρόπο ανοιχτό και διαφανή ούτως ώστε όλοι να εμπλακούν. Γιατί μας απογοήτευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άλλη μια φορά έφτιαξε ένα έγγραφο εργασίας για το προσωπικό τη, αλλά αυτό έγινε για άλλη μια φορά χωρί, να υπάρξει διαβούλευση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Επομένω, η κοινωνία των πολιτών ε, Πώ θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει. ακριβώ όπω γίνεται στι περιπτώσει ανακοινώσεων προ Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω, τώρα ήρθε η ώρα να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mr. Anley, what do you prefer? Ποιο τέλο πάντων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει. Ποιο Λορέντζο, ναι. Ναι, ναι, εγώ προσωπώ τη του περιβαλλον Περιβάλλον. Έχουμε διάφορε ερωτήσει, αλλά πρώτα-πρώτα να απαντήσω στον κύριο Ζαντό που είναι ο εισηγητή ε, και σχέση για την ε, Ινδονησία. Συμφωνώ μαζί του. Ναι, προσπαθούμε να πετύχουμε το στόχο μας και αλλά βέβαια είχαμε μόνο 5% των προϊόντων και είπαμε ότι όχι θα θέλουμε να πετύχουμε, δεν υπάρχει αξιοπία σε αυτό, οπότε το ξανασκεφτήκαμε και είπαμε να γίνουν όλες οι αλλαγές για τα έπιπλα και ε, πριν από ένα μήνα είχαμε μια συνεδρίαση, ήρθαν 25 Ινδονήσοι, τρεις εξατών ήταν από, ε, από την των πολιτών ή τα Υπουργεία και όλοι αυτοί ε, είπαν ότι θέλουν να τα συμφωνήσουμε και να δεσμευτούν. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία γιατί καλύπτουμε 100% των ε, σχετικών δραστηριοτήτων ακόμα και άσχετη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι θέμα αξιοπιστίας τους, το ξέρουν. Οπότε άμα ξαφνικά εδώ πέρα υπάρξει ένα ύποπτο φορτίο που θα φτάσει, όλα καταραίουν. Άρα συμφέρει και αυτούς και εμάς να εξασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Οπότε εμείς ε, στη γενική μας διεύθυνση ε, έχουμε δεσμευτεί και βέβαια η κοινωνία των πολιτών και η συμμετοχή της θεωρούμε ότι είναι εγγύηση επιτυχίας. Οπότε έχουμε συνεργαστεί αποδοτικά με τα κράτη-μέλη και ε, μπορώ να σας αναφέρω τις υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο που μας βοηθούν σημαντικά. Πάμε τώρα στις ερωτήσεις που αναφέρθηκαν όσον αφορά τον κανονισμό. Η απάντηση είναι καταφατική, ναι προβλέπονται κυρώσεις και το κάθε κράτος μέλος έχει ορίσει ακριβώς τι κυρώσεις θα επιβάλλονται. Έχουν ήδη ε, κάποιες περιπτώσεις επισύρει τέτοιες ποινές και έχουμε επίσης ε, επιθεωρητές από Σλοβενία και Σουηδία και αυτοί οι επιθεωρητές προσπαθούν στους εταίρους μας να α, τους δώσουν να καταλάβουν τι ισχύει, ότι υπάρχουν κυρώσεις. Θεωρούμε ότι οι σαλασσόμενοι πρόκειται να πάρουν το μήνυμα. Όχι, όχι, συμμετέχει στα του κανονισμού ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει πρόβλημα να πω στη γραμματεία σας ε, τις πληροφορίες που έχω. Να σου πω για τις δίκες που έχουν γίνει στα κράτη-μέλη, για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κλπ. Ναι, η υλοποίηση είναι κάτι το δύσκολο. Όπως είπαμε και στην εισήγησή μας, ε, συνεργαζόμαστε, ε, υπάρχει αλληλοβοήθεια, υπάρχει μετάδοση της πείρα για αυτά τα χρόνια και οπότε έχουμε θετικά αποτελέσματα σε μερικέ ε, περιπτώσεις, θα πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, ακριβώς όπως θα θέλατε κι εσείς να υπάρξει συνεργασία όσο γίνεται περισσότερο. Τελικά όμως θα πρέπει να είναι κανεί ε, αποφασισμένος να επιβάλλει αυτό που προβλέπεται. Επίση είπαμε ότι θα μην υπάρχει δυσανλογία, αλλά εάν κανείς είναι συναλλασσόμενος θα πρέπει να δει το θέμα της νομιμότητας της ξυλίας γιατί αν αρχίσει κανείς να ανακατεύει ε, τις πηγές προμήθειας των προϊόντων ε, τότε μπορεί κάποιοι από την πηγή, κάποιος από τους προμηθευτές να είναι παράνομος. Επομένως υπάρχει ακόμη περισσότερο κίνητρο να εξασφαλιστεί το ότι όλες οι πηγές είναι καθαρές και νόμιμες. Επίσης, αναφέρθηκε το ζήτημα της ε, συνέπειας. Όταν εγώ μίλησα για συνέπεια, αναφερόμουν ε, στο εύρος εφαρμογής του κανονισμού, ε, την ενδεχομένη αναθεώρηση. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η διαδικασία. Εμείς θα αξιολογήσουμε, θα διαβουλευτούμε, θα δούμε τις συνέπειες των μεταβολών, αλλά Βεβαίως και η αξιολόγηση μας έδειξε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα. Επίσης, βλέπουμε πόσο όλα αυτά σχετίζονται με την αποψήλωση των δασών. Όλα αυτά έχουμε αρχίσει να τα μελετάμε και να δούμε ποια είναι η πιο σωστή προσέγγιση. Περιμένουμε σχετικέ μελέτες και εκθέσεις. Ό,τι αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περάσει πρώτα από διαβούλευση με κρατημέλη και κοινωνία των πολιτών. Δεν θα γίνουν αυτά όλα κρυπτό και παραβήσω των Περλεμών. Όλα θα γίνουν με διαφάνεια. Ανοιχτά. Είναι περίπλοκα τα πράγματα όπως είπαν κάποιοι βουλευτές. Εδώ και δύο-τρία χρόνια είχαμε την πρώτη έκθεση που δημοσίευσαμε. οι αγορές των εμπορευμάτων είναι οι αποδέκτες αυτής όλης της δραστηριότητα. Καφές, κακάο και κλπ. Και όλα αυτά τώρα αναλύουμε και εξετάζουμε. Βεβαίω και είναι ενδιαφέρουσα αυτή η σχέση ε, με τα ορυκτά και τη σχέση ε, της ε, νομοθεσίας για τα ορυκτά με τον εν λόγω κανονισμό. Όταν μιλούμε για εμπορεύματα, υπάρχει πίεση από τα κράτη-μέλη. Άρα τα πράγματα εδώ περιπλέκονται. Ας πούμε το έλαιο, κοκοφίνικα, οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέξουμε. Okay, perhaps another uh, couple of questions to... Μια ομάδα από άλλε ερωτήσει, και θα κάνω και κάποιες παρατηρήσεις. Θα ε, εργαστούμε ως κλάστερ. Αυτό απαιτούν και οι αναπτυξιακοί στόχοι, SDGs. Ο αντιπρόεδρος Τίμερμαν συγγείται της όλης αυτής προσπάθειας. Θα περιμένουμε και τους επόμενους μήνες για να δούμε. Πώς μπορούμε να εργαστούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως ό,τι αφορά μέχρι τώρα το σχέδιο δράσης FLECT, θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο με τις υπηρεσίες. Εργαζόμαστε στενά με τη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Περιβάλλον και τη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ DEFCO και την DigiTrade και Grow πρέπει να τη συμπεριλάβουν σε αυτή την προσπάθεια και τα κράτη-μέλη όμως. Αυτή ίσως είναι και η μεγαλύτερη ανεπάρκεια μέχρι στιγμής. Δεν συνεργαζόμαστε αρκετά ακόμα τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Η αξιολόγηση κατέδειξε ότι δεν υπάρχει επαρκή συμμετοχή σε ό,τι αφορά λοιπόν το ίδιο το σχέδιο δράσης, με τις χώρες παραγωγούς και τις χώρες εταίρους, έχουμε το λεγόμενο φλέκτα ε, φασίλες στο πλαίσιο της ΦΑΟ. Και εκεί βλέπουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα στην τρίτη φάση του προγράμματος. Και αυτό ξεπερνά τις χώρες με τις οποίες έχουμε εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση και θέλουμε να στηρίξουμε και άλλες χώρες. Τι μας ανησυχεί όμως πολύ είναι ο μικρός ιδιωτικός τομέας που μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από αλλαγές σε ό,τι αφορά την νομιμότητα. Και γι' αυτό το περισσιακό έγγραφο εργασίας. Όπως είπα, ε, ουσιαστικά βλέπει τι έχει γίνει μέχρι τώρα, έγινε στο πλαίσιο του κανονισμού, του, πλαίσιο, του πακέτου, του σχετικού εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το μελετούν διάφορες υπηρεσίες. Όταν κυκλοφορήσει μέχρι τα τέλη του Ιουνίου θα μπορέσετε κι εσείς να το σχολιάσετε. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιολόγηση, την ανεξάρτητη αξιολόγηση, οι σύμβουλοι μας ε, είχαν ευρείες επαφές με τον ιδιωτικό τομέα, την κοινότητα των πολιτών, τις χώρες εταίρους. Ευχαριστώ. Thank you for ε, interesting... Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση και για τις παρουσιάσεις της Κομισιόν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη των τριών διαφορετικών επιτροπών. Εδώ ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο της μερισιάς διάταξης. Περιμένουμε δύο λεπτά να υποδεχθούμε τον Επίτροπο και έχουμε και ένα νέο θέμα στο πλαίσιο της Επιτροπής